Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου. Πρώτο θέμα, έγκριση της μεριζησίας διάταξη. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, να θεωρήσω ότι εγκρίνεται. Δεν βλέπω κανένα να θέλει να προσθέσει κάτι. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Τίποτα. Ωραία. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο, το 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 5 Νοεμβρίου 2018. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Περνάμε στο 4 τώρα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρώτο θέμα, εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Ε, do you point of order? Yes, please. Point of order. Well, I'm not sure point of order. Σημείο προς ενημέρωση. Αναρωτιέμαι, είναι απαραίτητο να ψηφίζουμε στις 4 τη Δευτέρα το απόγευμα. Πραγματικά μιλάω για τον εαυτό μου. Έφυγα στη μία για να μπορέσω να έρθω εδώ να ψηφίσω. Ίσως θα ήταν καλύτερο να γίνει αργότερα η ψηφοφορία. Δεν περιμένω να αλλάξει ο κανονισμός για μένα, αλλά θα ήθελα να σκεφτείτε ότι θα έχουν κάποια άποψη και τα άλλα μέλη. Αν η πλειοψηφία βεβαίως δεν συμφωνεί, εντάξει. Ε, παιδιά, δεν μπορώ να αλλάξω αυτό. Αγαπητοί φίλοι, σε γενικές γραμμές, ο χρόνος μας ε, πιέζει. Δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα να συναντηθούμε την επόμενη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Αν θέλετε να το αλλάξουμε, να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Ε, εγώ θεώρησα ότι το καλύτερο ήταν να συναντηθούμε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες. Ενδεχομένως Μερικοί από εσά δεν ικανοποιήθηκαν με αυτή τη ε, λύση και πολλοί από εσά δεν θα είναι καθόλου ικανοποιημένοι αν ψηφίσουμε τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Πάρα πολλέ φορέ έχουμε διαμαρτυρίε. Όχι ψηφοφορία στο Στρασβούργο. Και είναι και τη τελευταία μα συνάντηση για φέτο. Τελειώσαμε. Σε, σου ζητώ συγγνώμη, Σόνο. Είχαμε ενώπιόν μα. Ε, δύο κακές επιλογές και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Okay. Ε, let us start then. Reuse of public sector. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Αναδιατύπωση. Ξεκινήσαμε καλά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ah, okay. And να κάνουμε έναν έλεγχο. Ωραία. Test vote είπε ο πρόεδρος και κατά λάθο είπε sex vote. Thank very much. okay. Ωραία, ευχαριστώ. Σχέδιο έκθεση εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Επαναδιατύπωση. Ο συνάδελφος ο Σιλικιώτης είναι ο εισηγητής. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές δεκτό. 1.51 λίμπε 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ίνκο 38. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1.55. 5, 4, 5, 3 Ταυτόσημες υπέρ, κατά, να ελέγξουμε. I close the vote. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2α. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2β υπέρ κατά γκρίνεται 7-2. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 25 υπέρ κατά Μισό λεπτό να το ελέγξουμε. Λίμπε 25. Λίμπε 25. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 159 αντί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 190 είναι 43 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 ναι, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά να το ελέγξουμε λίγο τροπολογία 33 πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 34. Λίμπε 30 και οι δύο μαζί υπέρ. Κατά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ένα 196 107 υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε. Πέρας πληροφορίας Εγκρίνεται. Περνάμε στην 199, ΙΜΚΟ 44, υπέρ, κατά. Μισό λεπτό να το ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 200 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 202 υπέρ, κατά, Αποχές να το ελέγξουμε. 202. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μισό λεπτό να το ελέγξουμε. 36. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 47 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ήμκο 47 ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και λίμπε 31 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 209 ΙΜΚΟ 48 λίμπε 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λίμπε 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2, 213 λίβε 37 249 49 υπέρ κατά <clears throat> αποχές απορρίπτεται 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.15 ΙΜΚΟ 50 ΛΥΠΗ 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 217 ΙΜΚΟ 51 ΛΥΠΗ 39 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 2.17 και ΙΜΚΟ 51 και ΛΥΠΗ 39 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 2.19, ΙΜΚΟ 52, ΛΥΜΠΕ 40, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, ΛΥΜΠΕ 41, υπέρ, κατά, αποχές. Α, μισό λεπτό, θα ψηφίζουμε. ΛΥΜΠΕ 41, υπέρ, κατά, Α, εγκρίνεται. 2, 220, ΛΥΜΠΕ 42, υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. 220 και λίμπε 42. Πέρες ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ήμκο 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 222 D, 223 D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίνκο 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίνκο 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 255 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 256 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 257 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά Μισό λεπτό να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 45. 45 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά σας παρακαλώ επί της τροπολογίας 46. Rejected. Rejected. 258. 258D υπέρ κατά Ας το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά να είμαστε σίγουροι Πέρας της ψηφοφορίας Απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κουλτ 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Με συγχωρείτε, μισό λεπτάκι. 261, ξεχάσαμε τη 261. Ψηφίζουμε επί της 261 μετά την ΙΜΚΟ 75 που εγκρίθηκε παρακάμπτουμε τη 260 και πάμε στη 261 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμκο 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 273 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κούλτ 17 υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 313 ΙΜΚΟ 88 υπέρ κατά Ας το ελέγξουμε καλύτερα, να είμαστε σίγουροι να μην γίνει λάθος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 313. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 318 υπέρ, κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 318, πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 319 ΙΜΚΟ 90 υπέρ κατά αποχές ας ψηφίσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ Πέρα της προφορίες. απορρίπτεται συμβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην 67 ΙΜΚΟ 6 ΛΥΜΠΕ 4 υπέρ κατά αποχές Ας το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Λίμπε 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε καλύτερα αυτό. Ψηφίστε παρακαλώ επί 5. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. Όχι, όχι, εγκρίνεται, εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. Ήταν σαφές. 9. 9. Υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 9. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τροπολογία 9. Όχι τη Λίμπε 9. Τροπολογία 9. Για αυτή ψηφίσαμε τώρα. Ξαναλέω. Και επαναλαμβάνω. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 9. Πέρασε τις φοβορίες. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 82 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84 λίμπε 11, ΙΜΚΟ 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική F, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 90 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 91 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 89 λίμπε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά Α το ελέγξουμε καλύτερα αυτό. Ψηφίστε σας παρακαλώ ηλεκτρονικά επί τη τροπολογία 104. 104 και η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε απορρίπτεται. Συμβαστική Ι υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Κουλτ 3 υπέρ κατά εγκρίνεται εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κουλτ 4 υπέρ κατά ας το ελέγξουμε καλύτερα αυτό ψηφίστε σας παρακαλώ ηλεκτρονικά επί της κουλτ 4 και η ψηφοφορία ολοκληρώνεται απορρίπτεται ΙΜΚΟ 22 υπέρ κατά Α πούμε ότι εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά αποχέ εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 128 γιατί δεν βλέπω τα χέρια σας. Ψηφίστε σας παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 129D, ΙΜΚΟ 27D υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, ΙΜΚΟ 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 20 υπέρ, κατά Ας το δούμε καλύτερα ηλεκτρονικά, να το επαληθεύσουμε λέω. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 133 ΙΜΚΟ 30 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά αποχές ας το ελέγξουμε. Ψηφίστε σας για την τροπολογία 25 ηλεκτρονικά με τις κάρτες σας. Πέρας απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλτ 6 υπέρ, κατά Ας το ελέγξουμε και αυτό καλύτερα. Ψηφίστε σας παρακαλώ επί της Κουλτ 6 και η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. Ήμκο 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 149, ΙΜΚΟ 36, Λίμπε 22 που ταυτίζονται υπέρ. Κατά... Α, α, ας το ελέγξουμε καλύτερα. Τρεις τροπολογίες που ταυτίζονται, η 149 είναι η πρώτη, ψηφίζουμε, πέρας, απορρίπτεται. Λίμπε 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 150 ήμικο 37 που ταυτίζονται υπέρ κατά ας τις ελέγξουμε αυτές τις δύο καλύτερα ηλεκτρονικά πέρας απορρίπτεται και πάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά σας παρακαλώ Ψηφίζεται. Ψηφίζεται. Και η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή και περνάμε στην πληροφορία για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων υπό το άρθρο 69 γάμα του ιστορικού οικονομισμού. Εσωτερ... ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα και η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίθηκε λοιπόν και η εντολή αυτή για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ξέρετε ότι οι διαπραγματεύσει θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό. Οπότε ήταν απαραίτητο να γίνει ψηφοφορία φέτος. Ζητώ συγγνώμη για αυτό. Αλλά ξέρετε ότι η σημερινή μα συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί από την αρχή αρχή της χρονιάς. Δεν ήταν κάτι που έγινε τελευταία στιγμή. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ε, ήθελα απλώ ε, να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδη συγητές, τους συνεργάτες τους και του ανθρώπου από το γραμματεία της ε, Επιτροπής ε, μας, της ΙΝΤΡΕ, για την πολύ στενή συνεργασία που είχαμε. Ήταν πολύ παραγωγική η συνεργασία μας και ελπίζω ότι μαζί με τη στήριξη τους με, μετά από ότι θα μπούμε πολύ δυνατά στους λόγου για να εκπροσωπήσουμε επικοδομητικά και δυναμικά την άποψη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και πάλι όλους για την άψογη συνεργασία που είχαμε για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στο επόμενο σημείο το 5 ψηφοφορία για τη θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τον προοπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων. Ο συνάδελφος Πέτερ Κορουμπάσεφ είναι ο εισηγητής μας και ξεκινάμε ευθύ αμέσω. 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 και 6 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία, να ελέγξουμε. 18. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 18. Καλή ιδέα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 για την αιτιολογική ε, σκέψη 16 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 για την ε, ενωσιακή συγχρηματοδότηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά... Ας το ελέγξουμε καλύτερα αυτό. Ψηφίστε σας παρακαλώ επί της τροπολογίας 27. Και ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά... Αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά... Αποχές, Ας το ελέγξουμε καλύτερα αυτό. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 30. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να το ελέγξουμε. Δεν είμαι σίγουρος. Ψηφίστε σας παρακαλώ επί 11 αγαπητοί φίλοι, και κλείνω την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ψηφίζετε, σας παρακαλώ, και σταματάτε να ψηφίζετε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Τεράστια υποστήριξη, πλειοψηφία μεγάλη. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνούμε τώρα στο επόμενο θέμα. Και αυτό έχει θέμα και με τον προπολογισμό και θα πρέπει να ψηφιστεί και πάλι στην Ολομέλεια. Όλα τα θέματα που άπτονται του προπολογισμού θα πρέπει να ψηφιστούν και στην Ολομέλεια, διότι δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω διαπραγματεύσει σε επίπεδο επιτροπή. Περνούμε στο επόμενο θέμα. Ευρωπαϊκό Μηχανισμό στον τομέα τη πυρηνική ασφάλεια που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονία Ανάπτυξη και Διεθνού Συνεργασία βάσει τη συνθήκη Ευρατών. Ο εισηγητή είναι ο συνάδελφο Βλαντιμίρο Ρούτσεβ. Τροπολογίες 19-22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Να σηκώνετε το χέρι σας, παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος, για να βλέπω τα αποτελέσματα. Πάση περιπτώσει, ηλεκτρονική επαλήθευση. Στο 26 αρχίζει ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία, απορρίπτεται 28. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 και 10 το δεύτερο μέρος από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Έχει καλώς. 57 και το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 10 παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Με ισοψηφία. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, Όχι. Τροπολογία 61, όχι συμβαστική. Διορθώνει ο πρόεδρος. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επελήθευση και πάλι. Της 68. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 69. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 69. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 71. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Τι ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση, διότι δεν βλέπω με σαφήνεια τι ψηφίσατε. 74 λοιπόν. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται βεβαίω. Σας παρακαλώ, σηκώνετε το χέρι σας. 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σαφές το αποτέλεσμα. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Την 17. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Uh, amendment 17. Ολογία 17. The vote. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 16 και 18. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 78. Υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 79. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 80. Υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επαλήθευση στην 80. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82. 19. 24 και 2. Από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 83 και 49 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, λέει ο Πρόεδρος. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση στην 83 και 49. Εντάξει. I close Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 μαζί με την 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 1 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική απελευθέρωση. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση στις 27. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση της 6. Αρχίζει λίγη η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά και 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 47 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση της 47 λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία το σχεδίο έκθεση έτσι όπως τροπολογήθηκε. Οραμαστική ψηφοφορία, αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στην εισηγητή. Πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Κύριε Πρόεδρε, στην προηγούμενη έκθεση για τον δημόσιο τομέα, η τροπολογία μου 232 δεν τέθηκε σε ψηφοφορία, αφορά το νέο άρθρο 5, τροπολογία 232, στην προηγούμενη έκθεση αναφέρομαι. Θα ελέγξει το θέμα αυτό η γραμματεία και θα επανέλθουμε μετά την επόμενη ψηφοφορία γιατί θα χρειαστούμε χρόνο. Συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά θα το ελέγξουμε ούτως ή άλλως. Περνούμε στο επόμενο θέμα. Θέσπιση προγράμματο για την ενιαία αγορά, ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων και τι ευρωπαϊκέ στατιστικέ. τρία γνωμοδότηση η αντιπρόεδρο Πατρίτσια Τόγια. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση της 22. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Ε, με συγχωρείτε, 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση του 156. Απορρίπτεται. 157. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ. Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. And I close Έληξη ψηφοφορία και απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 26. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 171. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 189 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση της 189 λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές Πάλι δεν σηκώνεται το χέρι. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται. 190 και 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 44 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 213 υπέρ κα, ηλεκτρονική επαλήθευση της 213. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ ηλεκτρονική υπαλήθευση 47 λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται η συμβιβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 218 εγκρίνεται, 219 υπέρ, κατά, ηλεκτρονική επελήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 223 υπέρ κατά αελικρονική επαλήθευση του 223. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 28 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1, 1, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται 61 υπέρ κατά ηλεκτρονική επελήθευση της 61 παραλαμβάνει πρόεδρος λίγη η ψηφοφορία απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 64 Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 75 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 89 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 94 ε, υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται, 95 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, απορρίπτεται, συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 106 υπέρ κατά εγκρίνεται, 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ε, συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 126 υπέρ κατά Επιτέλους. 126 ηλεκτρονική επαλήθευση. And I close the vote. Is rejected. One... Απορρίπτεται. 130. Υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 130. Ναι, ναι, 130 διορθώνει ο πρόεδρος. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 131. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Του 131. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 143 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται. 144. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 145. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται 146 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση της 146 λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται και τώρα περνούμε στην ε, τελική ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει η ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία με συντριπτική πλειοψηφία και συγχαρητήρια στην συγκίτρια εγκρίθηκε. Και τώρα γυρίζουμε πάλι πίσω. Παρακαλώ. Παίρνω το λόγο για να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους και τους χιώδεις ε, για τη δουλειά που έκαναν. Πήρα όμως το λόγο για να πω το εξή. Από ό,τι ακούσαμε η Επιτροπή ΙΝΚΟ, στην οποία θα καταλήξει η δουλειά που κάναμε, δεν είναι ιδιαίτερα υπέρα Προσπαθήσαμε να κάνουμε μία δουλειά ιδιαίτερα ανοιχτή που συμπεριλάμβανε πολλές ε, επιχειρήσεις. Η Ίνκα ε, προσπαθεί να είναι περιοριστική. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους που έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν μέσω των ε, ομάδων να κάνουν κάτι γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ αλλά στο τέλος θα αποδεκατιστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Πατρίτσια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα σωστό έλεγχο γιατί θα πρέπει να γίνει ως ψηφοφορία στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και μετά θα πρέπει να περάσει στην Ολομέλεια και η Ολομέλεια θα ψηφίσει από την αρχή τα πάντα. στην ΙΜΚΟ είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε χωρίς ψηφοφορία. Σε ευχαριστώ Πατρίτσια. Πολύ σημαντικό αυτό. Περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Νεοκλή Σιλικιώτη, του συναδέλφου. Παρατήρηση του συναδέλφου είναι ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην τροπολογία 2.32, 2.32, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θα πρέπει να την ψηφίσουμε. Έχετε δίκιο. Μιλάμε για την έκθεση του κυρίου Σιλικιώτη. Εκ νέου χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Βρέστε το παρακαλώ. «2.32 ΙΜΚΟ 61 πριν από αυτό και μετά συμβαστική 9. Ψηφίζουμε τη 2-3-2. 2-3-2. Τροπολογία που υπέβαλε η κυρία Ρέντα. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Απορρίπτεται. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ρέντα ευχαριστώ που μας το θυμήσατε. Όντω είχε γίνει ένα λάθος. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Τα περισσότερα από τα θέματα θα υποβληθούν στην Ολομέλεια γιατί για θέματα δημοσιονομικά είναι απόλυτα αναγκαίο. Α, αν φεύγετε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε μία δεξίωση αν δεν σας ξαναδώ, καλά Χριστούγεννα. Ή επιστρέψτε σε μία ώρα. Μία, σε μία ώρα έχουμε την δεξίωση. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Το επόμενο θέμα Presentation of store στη παρουσίαση του ΣΤΟΑ. Παρουσίαση του ΣΤΟΑ λοιπόν για την τρισδιάστατη βιοεκτύπωση για ιατρικούς σκοπούς και για σκοπούς ενίσχυσης. Θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Η μελέτη μας παρέχει μια λεπτομερή ανασκόπηση των μελλοντικών εξελίσεων και των προοπτικών που παρουσιάζει η τρισδιάστατη βιοεκτύπωση και αναλύεται η επίπτωσή της. Μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα γιατί έχει κοινωνικές, ειδικές, δεοντολογικές και ε, κοινωνικές τυχές. Μπορείτε να δείτε στοιχεία για τη μελέτη αυτή διαδικτυακά στην ισοσελίδα του Κοινοβουλίου. Έχουμε τον φιλοξενούμενο διδική, τον κύριο Κρίστοφελ Κόνενα από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλσρούης. Παρακαλώ, κύριε Κόνεν, μπορείτε να περάσετε στην παρουσίαση και καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Well, if if anybody should leave immediately, it is even possible to say few words. For example, Madam Madam maybe Niebler or somebody else. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Δεν ξέρω. Θέλετε να φύγετε. Το θέμα είναι για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Στο τέλος της συνάντησης Έχουμε την Αντζέλικα Κανίμπελ που θα μας μιλήσει για το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ε, κατάλαβα ότι θα πρέπει να φύγετε, γι' αυτό αλλάξαμε τη σειρά. Λοιπόν, ένα-δυο λόγια για τον ε, ε, φορέα της ε, ε, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Κυρία Νίμπλερ, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά δεν θα σας κουράσω γιατί είχα την δυνατότητα και την προηγούμενη εβδομάδα να σας ενημερώσω για το θέμα της κυβερνοασφάλεια. Λοιπόν, την τελευταία εβδομάδα μετά τη συνεδρίασή μα, έγινε και ένα τριμερή διάλογο όπου καταφέραμε να προσεγγίσουμε ε, τα δύο άλλα θεσμικά όργανα σε αρκετά θέματα. Υπάρχουν όμως και κάποια ανοιχτά θέματα. Να σας ενημερώσω απλώς ότι τη Δευτέρα στο Στρασβούργο θα γίνει ο τελευταίος τριμερής διάλογος, αλλά είμαι βεβαία ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Ιδίως όσον αφορά την υποχρεωτική πιστοποίηση, τη διακυβέρνηση, εκεί είναι τα θέματα που θα χρειαστεί να συζητήσουμε και τα ευάλωτα σημεία. Αυτά τα τρία είναι τα θέματα που εκκρεμούν δεν έχει βρεθεί ακόμα συμφωνία, αλλά υπάρχει προθυμία και από τις τρεις πλευρές να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Δευτέρα βράδυ, τελευταίος τριμερός, τριμερής διάλογος. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Κατά τα άλλα δεν έχω κάτι να σας πω. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ ήταν το σημείο 13. Έχετε κάποια παρατήρηση. Όχι, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Περνάμε λοιπόν στο 8. Παρουσίαση του ΣΤΟΑ με θέμα τρισδιάστατη βιοκτύπωση για ιδρικούς σκοπούς και σκοπούς ενίσχυσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την μελέτη στόα μετά από ένα αίτημα του Ντάριο Ταμποράνο. Μαζί με τον ε, συνάδελφό μου θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που ενδεχομένω έχετε. Okay. It's a little bit, I'm sorry, it's a bit slow. Why is additive biomanufacturing or 3D printing a policy challenge? Το θέμα αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στις δύο και αυτό συμπεριλαμβάνει την χρήση πρόσθετων εφαρμογών, ε, βιολογικό δηλαδή υλικό, αλλά εξετάζουμε και κάθε είδους ε, ιατρικές χρήσεις. Ε, στα προσθετικά μέλη, για παράδειγμα, στο ιατρικό τομέα, Η τρισδιάστατη βιοεκτύπωση μπορεί να επιτρέψει την επιμέτρο προσαρμογή. Για παράδειγμα, προσθετικά μέλη στην οδοντιατρική μπορεί να επιτρέψει μια μείωση του κόστους, βελτίωση της ποιότητας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μη ιατρικούς σκοπούς. Είναι επίσης χρήσιμη για αποκέντρωση και αλλαγές στην αλυσίδα αξιών. Υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες για το μέλλον, συμπεριλαμβάνοντας ε, και τον μη ιατρικό τομέα, εφαρμογέ δηλαδή για σκοπούς ενίσχυσης. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές ε, ε τις διαδικασίες ε, για να ενισχύσουμε την απόδοση. Υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες, αλλά είναι ασαφές ακόμα για το πώς ε, αντιμετωπίζεται ε, οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και οι διοντολογικές. Εντοπίσαμε στη μελέτη, όπως μπορείτε να δείτε στο τελευταίο κεφάλαιο, τρία βασικά θέματα πολιτικής, ένα θέμα ρυθμιστικό, δεύτερο κατανομή των ωφελών και συμμετοχή του κοινού και καινοτομίε που προέρχονται από τους πολίτες. Για κάθε ε, θέμα έχει αναπτύξει, ε, η μελέτη έχει αναπτύξει δύο ξεχωριστού. κλάδους. Η πρώτη επιλογή εστιάζεται σε ρυθμιστικούς μηχανισμούς. Εδώ έχουμε δύο επιλογές και υπάρχει μία εξισορρόπηση μεταξύ της ειδικότητα των κανονισμών και της ταχύτητας. μπορείτε να δείτε ότι από την ε, μία πλευρά μας ενδιαφέρουν οι χρήστες και από την άλλη ορισμένες εφαρμογές. Λοιπόν, αυτός ο κανονισμός κινείται παράλληλα με τις καινοτομίες επιτυγχάνοντας μία ισορροπία. Α, μου είπα να μιλάω πιο αργά. Το άλλο θέμα αφορά την τύχη κατανομή των ωφελών. Εδώ υπάρχει μια εξισορρόπηση από την, ε, σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες εφαρμογές και την ανοιχτή καινοτόμο πολιτική. Υπάρχουν δύο αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρέ στον τομέα της τρισδιάστατης βιοεκτύπωσης. Αυτό που λέμε είναι ότι θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε περισσότερο εξειδικευμένες εφαρμογές και από την άλλη να έχουμε μία ευρύτερη προσέγγιση. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μία συζήτηση για τις ιατρικές συσκευές. Διαπιστώθηκε στην συζήτηση αυτή ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, πρέπει να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρξει ένα πιο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Περνάμε στο θέμα της συμμετοχής ε, του δημοσίου και της καινοτομίας ε, που προέρχονται από τους ε, πολίτες. Εδώ μπορείτε να κάνετε μία διάκριση σε ό,τι αφορά αυτούς που το συζητάν και που παρουσιάζουν διάφορες απόψεις σε ό,τι αφορά αυτές τις τεχνολογίες αποσκοπώντας τις μακρο, μακρόπνοες ιδέες χρήσης της τρισδιάστατης βιοκτήμωσης από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα κίνημα πολιτών που είναι καινοτόμοι και που αναπτύσσουν τεχνολογία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά από την άποψη της δημόσιας συζήτησης και της συμμετοχής του κοινού. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει νωρίς ο διάλογος προκειμένου να κατευναστούν οι προβληματισμοί. Και αυτό σε ό,τι αφορά τους τελικούς χρήστες. Αυτό θα ήταν χρήσιμο για ορισμένες αγορές θυλάκους, αλλά για να υπάρχει μια περαιτέρω εξέλιξη στην τεχνολογία. Και εδώ πάλι τίθεται το θέμα των εφαρμογών και, καθώς και θέματα ασφαλείας. να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση για να μπορέσει να γίνει κατανοητή, να γίνει κατανοητό το βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ε, δυναμικό, χρειάζεται μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Θα πρέπει κανείς λοιπόν να αποφασίσει που θέλει να εστιάσει την προσοχή της η Ευρώπη με βάση αυτές τις προσπάθειες εξισορρόπησης και ενώπιον του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Δεν θέλω και πάλι να αναφερθώ στο αυτό που συνήθως λέγεται ότι οι Αμερικανοί προηγούνται, αλλά θα πρέπει να πω ότι αυτό συμβαίνει στην αγορά και σε ό,τι αφορά την αλυσίδα αξίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σε ό,τι αφορά αυτές τις αντισταθμίσεις. Για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις εξελίξεις, προσπαθούμε να προωθήσουμε τη χρήση της βιοεκτύπωσης. Αυτές οι δραστηριότητες που προέρχονται από τους πολίτες ενδεχομένως θα πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής και στοχευμένης στήριξης. Όταν μιλάμε για ιατρικές συσκευές, αυτή η ιδέα της ανάπτυξής τους εκτός των εργαστηρίων πολύ συχνά αποτελεί πηγή προβληματισμών. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να πούμε ε, ότι θα μπορούσε να υπάρχει μία πρακτική ε, εφαρμογή αλλά παράλληλα να γίνεται και ένας πειραματισμός του χειμώνα συζητήσει μεταξύ των πολιτών. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη ε, βιοτεχνολογία, βιοκτύπωση στο μέλλον και η ανθρώπινη ενίσχυση, η επικοινωνία, ε, το κοινό είναι σε σημασίας προκειμένου να αποφευθεί ο ανώφελος και ή ο προβληματισμός. Τα, τα διάβασα πιο γρήγορα, τέλειωσα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ανέμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, ε, λέω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ νέα, αλλά και πολύ σημαντική στο μέλλον τεχνολογία. Κύριε Νίμπλερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση. Να σας πω την αλήθεια, δεν ήθελα να τοποθετηθώ για τι επιμέρου επιλογέ που υπάρχουν. Όμω, μπορείτε να μα ε, σκιαγραφίσετε ποια είναι η θέση, η εικόνα της Ευρώπης έναντι των άλλων ανταγωνισμών. Έχουμε κάποια πλεονεκτήματα, έχουμε κάποιο προβάδισμα, ε, ποια είναι, βρισκόμαστε ακόμα στην εφετηρία, ποια είναι η θέση των Αμερικάνων, ποια είναι η συγκριτική μα θέση σε σύγκριση με του Αμερικάνου ή με άλλου παίκτε ε, στο παγκόσμιο στερέωμα. Μπορείτε να μα δώσετε μια εικόνα. Πρόεδρο ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για τον καλεσμένο κείμενο μας. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γόνεν, Γιατί έχουμε προετοιμάσει και εμείς κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να αποτυχθούν πολύ ενδιαφέρουσες και για το δικό μας έργο εδώ στην Επιτροπή Ήτρε. Υψηλά πρότυπα για την βιοεκτύπωση, την τρισδιάστατη βιοεκτύπωση. Πώς μπορεί να κλείσει το κενό της νομοθεσίας που ισχύει σε διάφορες χώρες. Πώς μπορούμε να ερμονίσουμε τα κενά της νομοθεσίας μεταξύ των διαφορών χωρών, γιατί αυτό το θέμα της νομοθεσίας επί των προτύπων και των προδιαγραφών νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα. Δεύτερο, πώς μπορεί να ε, διαχειριστεί κανείς αυτή τη διαδικασία με εξειδικευμένες δεξιότητες. Νομίζω ότι η τρισδιάστατη βιοκτύπωση αποτελεί μια πάρα πολύ εξειδικευμένη ανθρώπινη δεξιότητα και αυτό μας ε, δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες για το πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί αυτή τη διαδικασία. Επίσης, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να χειριστεί το θέμα αυτό της βιοεκτύπωσης της ριάστατης με σκοπό να αποφευθεί η δημιουργία ολιγοπολίου. Νομικά ερωτήματα. Ποια νομικά ερωτήματα και θέματα αναδεικνύονται μέσω της τρισδιάστατης βιο, βιοεκτύπωσης. Γιατί νομίζω ότι αυτά τα θέματα μπορεί να είναι και πάρα πολύ περίπλοκα, θα μας απασχολήσουν στο μέλλον και υπάρχουν και ζητήματα ηθικής, αν θέλετε, δεοντολογικά, σχετικά με τη χρήση αυτής της νέας τεχνολογίας. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια πράγματα και για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικότερα ερωτήματα που ασχολούν το, το δικό μας έργο, το έργο της Επιτροπής Ήτρε. Αν μπορείτε να μας δώσετε και απαντήσεις, πραγματικά νομίζω ότι θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ στο έργο μας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά για εμάς. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Δεν βλέπω να ζητά κάποιος άλλος το λόγο, οπότε θα έλεγα να δώσουμε το λόγο στον προσκεκλημένο μας για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ για τα ενδιαφέροντα αυτά ερωτήματα. έχουμε προβάδισμα εναντί των άλλων ή έχουν οι άλλοι προβάδισμα εναντί ημών. Βλέπετε ότι η Ευρώπη, όπως και η ΙΠΑ και η Ιαπωνία, έχουν ε, προηγμένη τεχνολογία ιατρική και αντίστοιχη κατάσταση βεβαίως ισχύει και στον τομέα της βιοεκτύπωσης, της διάστατης και των βιοηλικών υπάρχουν έρευνες που συνεχίζονται σε διάφορους τομείς, σε διάφορα μέτωπα. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιο ηγέτη αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως πολλές εξειδικευμένε μικρές αγορές στι οποίε προχωράνε τα πράγματα. Αυτό βεβαίω αποτελεί και μεγάλη δυσκολία για τις κυβερνήσεις και για τις επιχειρήσει, προκειμένου να δημιουργήσουν ή να κατακτήσουν ή να εδρεώσουν μια ηγετική θέση γιατί το πεδίο είναι τεράστιο. Αντίστοιχε δυσκολίες ε, δημιουργούνται στο θέμα της νομοθετικής ρύθμισης όλη αυτή τη τεχνολογία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν, υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς στου οποίου οι εξελίξει είναι ραγδαίες ε, και υπάρχουν μια σειρά από ή υποτομεί όπου άνθρωποι ή ερευνητικά κέντρα προσπαθούν και βρίσκουν νέε εφαρμογέ για το BioAM, για αυτή τη μεταποίηση, αυτή την παρασκευή βιολογικών προσθέτων, τα οποία πρέπει να ε, ρυθμιστούν βεβαίως στο μέλλον νομοθετικά. Και γι' αυτό και καταλήξαμε σε αυτές τις επιλογές. Αν δείτε τις επιλογές, υπάρχουν μια σειρά αποτομής στο BioAM, αυτόν τον τομέα της τεχνολογίας που ε, αναδεικνύουν μια σειρά από νομικά ερωτήματα. Κάποια νομικά ερωτήματα είναι επίγοντα, είναι άμεσα και επιτακτικά και είναι να απαντηθούν και ε, ε, είναι και δύσκολο να απαντηθούν. Ένα από τα ερωτήματα από αυτά είναι ότι κάποια από αυτά τα προϊόντα ήδη χρησιμοποιούνται ως ιατρικές εφαρμογές και εντός, για παράδειγμα, του οργανισμού, του ανθρώπινου οργανισμού και ε, έχουν παρόμοιο αν θέλετε αποτέλεσμα και αντίκτυπο με τα φάρμακα, τα οποία ρυθμίζονται όμως νομοθετικά πάρα πολύ αυστηρά, χωρίς τα ίδια αυτά προϊόντα να ρυθμίζονται αντιστοίχως αυστηρά. Άμα δείτε τις εφαρμογές BioEM, δεν είναι πάντοτε σαφές που εμπίπτουν ε, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι συσκευές, είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα, είναι φάρμακα, είναι ουσίες δραστικές, είναι μη ανθρώπινες ουσίες, είναι βιολογικές ουσίες. υπάρχουν βιολογικές ε, εφαρμογές οι οποίες δημιουργούν ε, μη ανθρώπινο ιστό, για παράδειγμα, αυξητικό ε, ιστό. Υπάρχουν άλλες βιοφαρμογές οι οποίες ε, ε, δημιουργούν ανθρώπινο ιστό. Όλα αυτά δεν ρυθμίζονται ακόμα με ξεκάθαρο τρόπο στην νομοθεσία. Τρισδιάστατη βιοεκτύπωση. Εδώ ένα ερώτημα σημαντικό είναι τι κάνουμε. ποιος, τι ακριβώς πρέπει να ρυθμιστεί. Το υλικό, το λογισμικό, ο σχεδιασμός αυτών των προϊόντων. Όλα αυτά μαζί. Στο παράρτημα 2 της μελέτης μας ε, αναδεικνύεται ότι υπάρχουν ε, και φαίνεται ότι υπάρχουν μια σειρά από νομοθετήματα που ρυθμίζουν μεν το θέμα, χωρί όμω να συμβαδίζουν με τι τελευταίε επιστημονικέ και τεχνολογικέ εξελίξει. Εδώ είναι που έρχεται ο ρόλο Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει ένα σύνολο κανόνων για να καθοριστεί το πώ ακριβώ τελικά θα χρησιμοποιούνται, πώ θα κατασκευάζονται, πώ θα παρασκευάζονται, πώ θα χρησιμοποιούνται όλε αυτέ οι βιοεφαρμογέ, όλα αυτά τα βιοπροϊόντα. Και αυτό μπορεί και να απαντά και στο ερώτημα του κενού του νομοθετικού μεταξύ των διαφόρων χωρών. Αν δηλαδή θα μπορούσε ένα τέτοιο ενωσιακό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τις δικές τους νομοθεσίες. Αυτά για τα νομικά ερωτήματα. Ναι, νομίζω ότι ε, απαντήθηκαν τα περισσότερα ερωτήματα, αλλά θέλω να πω κάτι για το πρώτο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή η αγορά των ε, εφαρμογών υγείας δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη ακόμη. Βεβαίως υπάρχουν προβλέψεις ε, που είναι πάρα πολύ ενθουσιώδεις και αισιόδοξε. Αυτή τη στιγμή ε, θα μπορούσα να πω ότι συμβαδίζουμε ε, στον ένα στον άλλο βαθμό με τις αμερικανικές ε, επιχειρήσεις. Όμως αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο για το μέλλον. Μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν. Και εδώ θέλω να ε, τονίσω αυτό που είπε και ο συνάδελφος. Υπάρχει, είναι μια τεχνολογία διατομεακή αν θέλετε, διεπιστημονική. Υπάρχουν μια σειρά από πτυχές που εμπλέκονται με διαφορετικό, με άνισο τρόπο αν θέλετε μέσα στην, στην, στη διαδικασία παρασκευής αυτών των προϊόντων. Ε, γι' αυτό και πολλά πράγματα είναι άγνωστα. Υπάρχουν ε, βιοεφαρμογέ που κατευθύνονται και προορίζονται για τον ιατρικό τομέα, υπάρχουν όμως και αντίστοιχε εφαρμογέ που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και αυτό είναι προβληματικό και επικίνδυνο σε τομεί εκτός τη ιατρικής. Τι γίνεται λοιπόν εκτός τη ιατρική Εδώ υπάρχουν πάντοτε κάποιοι hacker ή κάποιοι επιστήμονε παρείε οι οποίοι ε, ε, επιδίδονται σε έρευνες ή σε δοκιμές, σε πειράματα με τέτοιες και αυτά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά πράγματα. Ε, ταυτόχρονα όμως αυτές οι βιοφαρμογές γίν, βρίσκονται, είναι, είναι ήδη μια πραγματικότητα και είναι πολύ ελπιδοφόρες. Δηλαδή εκεί που, όπου οι ίδιοι οι πολίτες μπαίνουν επικεφαλής αυτής της διαδικασίας, της ερευνητικής αν θέλετε και των δοκιμών, και εκεί ανοίγονται διάφοροι ορίζοντες που αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Επίσης, τέθηκαν ερωτήματα για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα υψηλού κόστους ή από τις επιλογές μας τι, τι κόστος προκύπτει. Εμείς είμαστε υπέρ της ανοιχτής ε, ε καινοτομίας ε, και της χρηματοδότησης βεβαίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με όλα τα προβλήματα που αυτά, αυτή η διαδικασία έχει, αλλά νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια πανευρωπαϊκή τυποποίηση. και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και μια συνάντηση ενός σχετικού δικτύου όπου οι εμπλεκόμενοι και οι συμμετέχοντες του δικτύου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλοι διάφοροι φορείς που ασχολούνται με αυτή τη διαδικασία και αυτή τη τεχνολογία ζήτησαν και ήδη αυτόν τον πιο συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ρυθμιστικού πλησίου γιατί θα ωφελήσει συνολικά. είναι γεγονός ότι αν αφαιθεί η όλη διαδικασία στα χέρια των επιμέρους ε, φορέων τότε μπορεί να δημιουργηθούν προβληματικές ε, καταστάσεις. Και τέλος για τις ανθρώπινες ε, δεξιότητες. Νομίζω ότι αυτό σχετίζεται και με την απώλεια θέσεων εργασία. Εδώ επισημαίνουμε και το ίδιο είπε και ο Ευρωβουλευτή Τεμποράνο, ότι το εξετάσαμε αυτό το θέμα ιδίως υπό την οπτική της οδοντιατρικής ε, η ανοιχτή καινοτομία, η έρευνα πρέπει να συμπεριλάβει ιδίω του επαγγελματίε, όχι μόνο του πανεπιστημιακού ή τι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται, αλλά του επαγγελματίε, του επιστήμονε. Γιατί αυτοί είναι πραγματικά εκείνοι που γνωρίζουν σε ποιο βαθμό μπορεί να ωφελήσουν αυτέ οι τεχνολογίε στου ανθρώπου, πώ μπορεί ένα άνθρωπο πραγματικά να, χρησιμε... να του χρησιμεύσουν αυτέ οι. Ε, οι τεχνολογίες, δηλαδή να μην μιλάμε μόνο με επιμελητήρια ή συνδικάτα ή οργανώσει επαγγελματιών, ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ η Ευρώπη πραγματικά βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της ε, διαδικασίας στον κόσμο του να φέρει τους πολίτες της όσο το δυνατόν στο επίκεντρο της προσοχής της προκειμένου να δημιουργηθούν προϊόντα τα οποία πραγματικά θα ανταποκρίνονται και στις ανάγκες των πολιτών της. Ευχαριστώ πολύ. Ζητά κανένας άλλος συνάδελφος το λόγο. Θέλει να κάνει κανείς και μια συμπληρωματική ερώτηση. So, thank you very much. Βλέπω ότι δεν ζητά κανεί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και είναι πολύ σημαντικά να γίνουμε πρωτοπόροι στο θέμα αυτό, να μην είμαστε στην ουρά. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να προχωρούμε πάντα μπροστά. Πολύ καλά συνοψίσατε το όλο θέμα. Η Επιτροπή θέλει να πει κάτι. Ευχαρίστως. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απλώς θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και μια ερώτηση. Θα ήθελα να πω ότι γενικά ο όρος bio, το βίο είναι κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθος. Δεδομένου ότι αν μιλούμε για bio εκτύπωση, ίσως μπορεί να οδηγήσει στην εκτύπωση κιτάρων και αυτό βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Το λέγω απλώς ως σχόλιο. Κατά τα άλλα μας πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετικές και εμπεριστατωμένες οι εκθέσεις σας Απλώς ήθελα να θέσω στη συζήτηση το σχόλιο αυτό. Και υπόψη Παρακαλώ, θέλετε να απαντήσετε. Βλέπω ακριβώς τι εννοείτε. Αυτού του είδους τα σχέδια συμπεριλαμβάνουν πάρα πολύ πολλά θέματα, τον βίο εκτύπωση, και το θέμα που αναφέρεται, τους ε, τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται, αλλά βεβαίως μπορεί κανείς να κάνει και διαχωρισμό και διαφοροποίηση μεταξύ της, ε, των ιατρικών χρήσεων που χρησιμοποιείται το πρόθεμα bio και για άλλες χρήσεις. Και βεβαίως υπάρχουν και οι άλλες χρήσεις, όπως είπε και ο συνάδελφος, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αυτοί που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις το λαμβάνουν υπόψη. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το 9 και το 10. Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αναδιατύπωση και κοινή κανόνες εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για θέματα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά και αφορούν, αφορούν το σχεδιασμό της εσωτερικής αγοράς και την ε, καθαρές, ε, καθαρά πακέτα ενέργειας. Ο συνάδελφος κύριος Κάρινς, ο οποίος είναι εισηγητής, δεν μπορεί να είναι εδώ, αλλά μου έστειλε κάποιες παρατηρήσεις. Πριν από δύο εβδομάδες έλαβαν χώρα ε, ο τρίτος και ο τέταρτος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών και συζητήθηκαν τα πακέτα σχεδιασμού της ηλεκτρικής ενέργειας και όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τα ε, ε όργανα που χρησιμοποιούνται, τα ε, στις οικολογικούς την ασφάλεια του εφοδιασμού, την διακυβέρνηση, κανόνες, καταναλωτές, τιμές και πρέπει να πω ότι γενικά επιτεύχθηκε πολύ καλή πρόοδος και έγιναν και συμβιβαστικέ λύσεις. Κάποια σημαντικά θέματα όπως ε, το θέμα της τιμολόγησης ε, και κάποια θέματα χρησιμοποίηση κάποιων ενεργειών παραμένουν ε, εκρεμεί. Αυτά μπορώ να σας πω. Εάν θέλετε συμπληρωματικές πληροφορίες, είναι στη διάθεσή σας ο εισηγητής. Ε, στην περίπτωση του κανονισμού πρέπει να πω ότι στα θεσμικά όργανα επιτεύχθηκε συμφωνία όσον αφορά τις γενικότερες διατάξεις των φορέων για την δύναμη της ενέργειας. Θα υπάρξουν ε, για τα θέματα αυτά περιφερειακά συντονιστικά κέντρα και αυτά τα θέματα είναι θέματα για τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να μπορεί επίσης να παίρνει Αυτό είναι ε, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Στον τέταρτο λοιπόν αυτό διάλογο μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων πρέπει να πω ότι επιτεύθηκαν συμφωνίες που μας επιτρέπουν να μειώσουμε σε πολύ σημαντικά θέματα που παραμένουν εκκρεμή ακόμη τις ε, διαφορές που υπήρχαν. Πρέπει να πω ότι επόμενος κοινός διάλογο μεταξύ των τριών κρατών μελών για τον σχεδιασμό της ηλεκτρικής αγοράς προβλέπεται στις 5 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα, πριν από τα Χριστούγεννα λοιπόν. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί τα τρία θεσμικά όργανα είμαστε ανοιχτά και ε, διατεθειμένα να συνεχίσουμε τον διάλογο μεταξύ ημών και στις 6 Δεκεμβρίου αν χρειαστεί για τον κανονισμό και την οδηγία που παραμένουν ακόμη εκκρεμή σε κάποια θέματα. Υπάρχουν ερωτήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι προφανώς αυτό είναι το τελευταίο μέρος ενός πολύπλοκου ε, θέματος. Έχουμε φτάσει σχεδόν αρχές Δεκεμβρίου, ίσως δεν έχουμε χρόνο. Δεύτερον, ξέρετε, διότι για πολλά θέματα έχουμε συνεργαστεί, ότι θα ήθελα να μην ε, χαθεί τίποτε όσον αφορά το πακέτο και την νομοθεσία για πολύ καθαρή ενέργεια προς όφελος όλων των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω συμβαίνει κάτι τέτοιο γιατί συζητάμε όλα τα θέματα και σε γενικές γραμμές υπογραμμίζουμε τα θέματα που είναι καθοριστική σημασίας για το Κοινοβούλιο. Έχετε δίκιο ότι ο χρόνος πιέζει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάστηκε να ψηφίσουμε απόψε. Ακόμα και αν αυτό δεν εξυπηρετούσε πάρα πολύ πολλούς συναδέλφους. Ήταν απαραίτητο να γίνει η ψηφοφορία. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε περάσει στο 11. Το θέμα 11 είναι παρεμφερές ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο συγητής, ο συνάδελφος Πέτερσεν, μου έστειλε επίσης μερικά πληροφοριακά στοιχεία. ετοιμότητα αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρική ενέργεια έκανα λάθο ο συνάδελφος Φλάβιο Ζαντονάτο. Ευτυχώς είσαι εδώ Φλάβιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, βιώσαμε μαζί αυτή την περιπέτεια στις 22 Νοεμβρίου. Τα τρία μέρη κατέληξαν σε μία συμφωνία την πρόταση κανονισμού για την ετοιμότητα αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό υπήρξε αποτέλεσμα του τρίτου τριμερούς διαλόγου όπου δεν έλειψαν στιγμές έντασης με την Προεδρία Το ε, τέλος. Το κείμενο οδήγησε σε μία συμφωνία και επέτρεψε στις αρχές χρόνους πολύ πιο παρατεταμένους. 30 γιατί 24 μήνες που ήταν αυτή που ζήτησε το Κοινοβούλιο για την εισαγωγή των πρώτων προγραμμάτων για τον ε, κίνδυνο. Ένα αποτέλεσμα θα έλεγα σημαντικό γιατί το κείμενο στην ουσία βγαίνει μετά από τις συζητήσει αυτές ενδυναμωμένο. Το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να μειώσει την περιφερειακή διάσταση και ο πρόεδρος ε, δεν κατάφερε να περιθωριοποιήσει το Άστσερ και να ε, επανεξεταστούν τα RCC και ο αποκλεισμό του από τη διαδικασία αξιολόγηση του κινδύνου και από τη σύνταξη των διαφόρων προγραμμάτων. Με λίγα λόγια, εξασφαλίσαμε την εφαρμογή τη αρχή τη αλληλεγγύη, που είναι βασικό άξονα αυτή τη πρόταση κανονισμού, με ουσιαστικό τρόπο, με τα απαραίτητα μέτρα ευρωπαϊκής και περιφερειακής εκ των προτέρων αξιολόγησης. Η ε, πολιτική σημασία μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα και άλλων να το σχέ προς την κατεύθυνση που θέλει το Κοινοβούλιο. Δεσμεύσαμε τον Συμβούλιο και αυτό πιστεύω ότι αποτελεί κάτι πολύ θετικό για μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολλούς. Επιτρέψα μου να επικεντρωθώ σε έναν, στον πρόεδρο Μπούζεκα, γιατί συνέβαλε καθοριστικά με την εμπειρία του και με την ε, δυνατότητα, την διαπραγματευτική του ικανότητα στην ισορροπία των, του τελικού κειμένου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη γραμματεία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Uh, Ευχαριστώ πολύ Φλάβιο. Πραγματικά μεγάλη επιτυχία. Επιτυχία πρωτίστως δική σου. Γιατί όλες οι διαπραγματεύσεις εξαρτήθηκαν από την προετοιμασία που έκανε εσύ. Εσύ εκπροσώπησες όλο το Κοινοβούλιο. μα μας υποστήριξε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο επέδειξε μία αρκετά ανοιχτή στάση. Καταρχάς, ε, θερμά συγχαρητήρια σε σένα, Πλάθιο Τζαντονάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Γιατί ήταν πολύ σημαντικό να πάρεις το λόγο και να πεις κάτι προς όλους μας. Έχουμε τέσσερις νομοθετικές προτάσεις στο δεύτερο μέρος του πακέτου καθαρής ενέργειας. Το δεύτερο μέρος τελείωσε πριν από ε, μερικούς μήνες και τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος, τέσσερες ε, νομοθετικές προτάσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει κάποια ερώτηση για τον συνάδελφο της Όχι, ωραία. Επιτρέψτε μου να πω ότι το τέταρτο, η τέταρτη νομοθετική πρόταση αφορά την Acer, τον φορέα για τη συνεργασία των ρυθμιστών ενέργειας, ο εισηγητής είναι ο κύριος Πέτερσεν που μου έστειλε ένα μικρό σημείωμα το οποίο είναι στη διάθεσή σας. Στην αρχή έγιναν τρεις τριμερείς διάλογοι. Καταλήξαμε σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα θέματα, όπως για παράδειγμα η πρόσβαση των ρυθμιστικών φορέων στην πληροφόρηση επόμενος τριμερής διάλογος θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Ελπίζουμε να είναι το τελευταίο, και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα. Έχουμε ακόμα επιτάπητο σημαντικά θέματα. Η ικανότητα του ΆΣΕΡ, της ρυθμιστικής αρχής, να παίρνει αποφάσεις σχετικά με περιφερειακά κέντρα συντονισμού. Υπάρχουν, ε, υπήρξαν ορισμένες αντιστάσεις από ορισμένα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο ε, έχουν αντιρρήσει στο να αποκτήσει τέτοιες δυνατότητες το Acer. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν δεν θα, είναι βραδίες και θα είναι δύσκολες. Αυτό το έχει υπόψη του εισηγητής. Ο, ο ρόλος του διευθυντή σε σχέση με το διοικητικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η θέση του Συμβουλίου είναι ξεκάθαρη. Θέλουμε έναν ισχυρό διευθυντή όσο γίνεται περισσότερο ανεξάρτητο που θα μπορέσει να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των ρυθμιστικών φορέων, τον ναι, Acer. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό φάκελο που αφορά το μέλλον της ηλεκτρικής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, αναφέρθηκα στα πιο σημαντικά θέματα. Παρόλα αυτά πιστεύουμε να ολοκληρωθούν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις στο Στρασβούργο στις 11 Δεκεμβρίου. Κάποιος θα ήθελε το λόγο αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν τέσσερις νομοθετικές προτάσεις που θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο για να μπορέσουν να γίνουν οι ε, περαιτέρω διαπραγματεύσεις υπό την ε, Προεδρία της ε, Ρουμανίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση. Κατά την άποψή Ψήσας, Ένα μέρος των διαπραγματεύσεων, ε, τα ΆΣΑΡ, εξαρτώνται από τους κανονισμούς στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πώς θα συνεχίσουμε όμως ε, σε περίπτωση που υπάρξει αποτυχία. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικά σενάρια αν κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους κανονισμούς. Μου έχετε απόλυτο δίκιο. Εξαρτάται τι θα αφήσουμε για τον τελευταίο τριμερή διάλογο ε, για τις 19 και 20 Δεκεμβρίου. Ε, ενδεχομένως θα είναι δυνατόν να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις μας για το ΕΣΕΡ. Αν όχι, θα είναι αναγκαίο να συναντηθούμε και πάλι στις 21 Δεκεμβρίου. Εγώ είμαι απόλυτα ανοιχτή το ενημέρωσα και το Συμβούλιο και την Επιτροπή, εξ ονόματος της Επιτροπής ε, Ήτρε, ενημέρωσα και τον εισηγητή βεβαίως, το ε, θα έρθω 19-20 Δεκεμβρίου, είναι πράσινη εβδομάδα, αλλά πράσινη εβδομάδα σημαίνει ότι είμαστε τιμοπόλεμοι. Δεν έχουν ε, ξεκινήσει οι διακοπές. Ως μέλη του Κοινοβουλίου δεν είμαστε σε περίοδο ε, διακοπών. Το θέμα είναι αν ε, είναι έτοιμο κανείς να έρθει τέσσερις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Για μένα πρόκειται για ένα καθοριστικό θέμα. Θα πρέπει να τελειώσουμε το Δεκέμβριο. Συνάντησα με ε, προσώπου από την ε, Προεδρία της Ρουμανίας και της Αυστρίας και θα ήταν καλύτερο και από την άποψη της Ρουμανίας, γιατί έχουν πολλά θέματα τάπιωτος. Καταρχάς θέματα δημοσιονομικά για τα επόμενα επτά χρόνια. Αυτά είναι θέματα που θα απασχολήσουν τη Ρουμανική Προεδρία από αυτή την άποψη. Λοιπόν, είναι απαραίτητο να τελειώσει αυτό το πακέτο καθαρής ενέργειας το Δεκέμβριο. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, έχετε δίκιο, δεν μπορούμε με το Acer ε, να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο, δίχως να ολοκληρωθεί το θέμα με την αγορά καθαρής ενέργειας. Κάποιο άλλος, το λόγο, όχι. Πράξη για την κυβερνοασφάλεια. 13. Μας ενημέρωσε ήδη η συνάδελφος πριν από μια ώρα. Δεν τέθηκαν ερωτήματα από τους ευρωβουλευτές, οπότε μπορούμε να περάσουμε στην, στο σχέδιο έκθεσης του Μύροσλαβ Πόχε προσαρμογή της οδηγίας 2012-27 για την ενεργειακή αποδοτικότητα και του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αυτή την ασυνήθιστη περίσταση. Το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει. Ο Μύροσλαφ Πόχα λοιπόν είναι ο εισηγητής μας στις 13 Νοεμβρίου η Κομισιόν υπέβαλε την σχετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και τη διακυβέρνηση, τον, κανονισμό μάλλον για τη ε, διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης για να καλύπτεται πλέον η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται δηλαδή για μια τεχνική προσαρμογή ε, σχετικά με την τελική ενεργειακή κατανάλωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η πραγματική κατάσταση μετά το Brexit. Δεν μας ε, επιτρέπει ο χρόνος λοιπόν να ε, πλατιάσουμε. Είναι απαραίτητο να ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή έως το Μάρτιο του 2019 ημερομηνία αποχώρησης της Βρετανίας. Και έτσι η Κομισιόν προσπά... Ε, αποφάσισε να προτείνει την, ε, να ακολουθηθεί μια διαδικασία επιταχυμένη και αυτό αφορά η έκθεση του κυρίου Μύροσλαβ Πόχε. Ο εισηγητής μας ε, έχει ζητήσει από την κυρία Τερέζα Γκρίφιν να τον υποκαταστήσει σήμερα και να μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ Τζέζι. Πραγματικά τι ηρωνία να σας ε, παρουσιάζω εγώ αυτό το θέμα. Ξέρετε ότι εγώ ήθελα να παραμείνουμε, ούτε θεωρώ ότι το πράγμα έχει τελειώσει. Η δε ψηφοφορία θα γίνει τα γενέθλιά μου. Ε, ελπίζω να είναι ένα θετικό δώρο, ένα ωραίο δώρο για μένα. Καταρχά, λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Μύροσλαβ που δεν μπόρεσε να, να παραστεί σήμερα εδώ. Μιλούμε για την προσαρμογή της οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα από τα, από τις, μία από τι ε, οχτώ νομοθετικέ πράξει της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να τροποποιηθεί. Πρόκειται για έναν επαναπολογισμό σε τεχνικό επίπεδο των καταναλώσεων και των εξοικονομήσεων ενέργεια. Τον προηγούμενο μήνα η Κομισιόν κατέληξε σε τελική συμφωνία με το Συμβούλιο που ορίζει 32,5% μείωση της ε, κατανάλωσης έως το 2030 στο ζήτημα της πρωταρχικής και της δευτερογενούς ενεργειακής κατανάλωσης. Η κατανάλωση στην Ευρώπη των 28 δεν θα πρέπει να ε, υπερβαίνει τα, τα 9,65 MTOE το 2020. Μετά την αφαίρεση των προβλέψεων ενεργειακή κατανάλωση του Ηνωμένου Βασιλείου μιλάμε πλέον για 1130 ε, και 948 ε, μονάδες. Ε, ο εισηγητή έχει κάνει κάποιε καθαρά τεχνικέ τροποποίησει, ιδίω όσον αφορά το στόχο 2. Το 32,5% να αφορά και την πρωτογενή και την τελική κατανάλωση και περαιτέρω προσδιορίζει ε, κάποια στοιχεία της ε, νομοθεσίας. Τέλος, η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από 20 σε 30 μέρες, γιατί στα 20, ε, στις 20 μέρες ενδεχομένως να μην είχαμε χρόνο για τις 29 Μαρτίου ε, του 2019, την ημερομηνία που προβλέπεται να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εισηγητή θεωρεί ότι η, κατάσταση θα, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ομαλά. Το Συμβουλίο ίδιο έχει πει ότι δεν θα, ε, προσφέρει, δεν θα φέρει προσκόμματα. Αν και ολοκληρώνοντα, θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω την ελπίδα μου ότι όλα αυτά τελικά δεν θα χρειαστούν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Είναι μια παράδοξη αυτή η κατάσταση. Το ότι σας ζητάμε εσάς, σε την κατάσταση των αδέλφων μας, την έκθεση αυτή. Αλλά γνωρίζουμε ποια είναι η θέση σας γενικότερα για αυτά τα οποία συμβαίνουν μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου αλλά σεβόμεθα τις δημοκρατικές αποφάσεις, γιατί δεν έχουμε άλλη δυνατότητα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. πάση περιπτώσει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση εξ ονόματος του Μυροσλάβ Πόχε. Και ήταν πολύ σαφής. Θα ήθελα ίσως να ρωτήσω την ε, Κομισιό, αν θέλει να κάνει κανένα σχόλιο. Κύριε Χότσον, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο μετά την παρουσίαση της κυρίας Γκρίφιν. Βεβαίως έκανε την παρουσίαση εκ μέρους του κυρίου Μυροσλάβ. Ευχαριστώ ίσως. Και... Απλώ τρία παρατηρήσει θα ήθελα να κάνω. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώ και το Συμβούλιο για την ταχύτητα με την οποία εξέτασαν αυτό το τεχνικό φάκελο. Τώρα, επί του περιεχομένου, δεν έχω να προσθέσω τίποτε στην έκθεση και κ. Πόχε και την παρουσίαση της κυρίας Τερέζα. Συμφωνούμε, βλέπουμε ποια είναι η σημασία των τεχνικών ε, ε, τροπολογιών και το πέμπτη για την ε, πολύ σωστή επιλογή που έγινε για την διαφοροποίηση αυτής της προθεσμίας 20-30 μέρες. Νομίζω ότι όλα θα γίνουν έγκαιρα λαμβάνοντας υπόψη το θέμα αυτό. Ευχαριστώ σας, ευχαριστούμε Τερέζα, θέλεις τώρα να πεις κάτι εκ μέρους του Μυροσλάβ. Απλώς ότι προφανώς προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε ε, λύση ενδεχομένως, τα παίρνουμε πολύ σοβαρά τα πράγματα. Χαιρόμαστε που το 32,5% στόχος αυτός είναι ένας στόχος που θα μπορούσε να ήταν υψηλότερος, αλλά χαιρόμαστε ότι θα μπορέσουμε να τον επιτύχουμε. Εγώ θα ήθελα 40% ε, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ πάλι Τζέσι βλέπεις πόσο εύκολα και με την δική σου ηγεσία όλες οι πολιτικές ομάδες κατέληξαν σε συνένεση προς τον των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή είναι η ομορφιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό νομίζω ότι μπορεί να με κάνει να πω ότι θα έπρεπε και για αυτό το λόγο να παραμείνει μεταξύ των 28 το Ηνωμένο Βασίλειο. Συμφωνώ μαζί σου, Τερέζα, συγκεκριμένη περίπτωση. Συμπερασματικά θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η Δεκεμβρίου 2018 και μετά θα ψηφίσουμε στις 14 στην Ήτρε και θα επιβεβαιωθεί για αργότερα η ψήφιση της έκθεσης αυτής στην Ολομέλεια. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου και την παρουσίαση Τερέζα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ήσουν εδώ και παρουσία στην έκθεση που είναι ίσως ε, κάτι το... Όχι χρήσιμο αυτό που θα πω, για να μην επαναλαμβάνουμε, αλλά κρίμα που χρειάζεται να λύνουμε τέτοιου είδους προβλήματα και ξέρουμε ότι όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι τέλος Ματιού. Αγαπητοί συνάδελφοι, στα διάφορα, συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να πω ότι Έχουμε λίγο χρόνο πριν από την, ε, τον εορτασμό τον Χριστουγεννιάτικο. που θα αρχίσει στις 8 και και στις, στις 6 και 4 και στις 6.30 θα έρθουν και δύο επίτροποι. Στο Γιάν, στην πρασρή του τρίτου ορόφου Εκεί θα γίνει η δεξίωσή μας Χριστούγεννιάτικη. Πολύ ωραίο μέρος. Σας καλώ λοιπόν στις 6 και 4, δηλαδή σε μισή ώρα από τώρα. Αλλά μην αργήσετε, μην αργήσετε πολύ. Δεν πρέπει να αρχίσουμε, είπαμε. Σε 6.30 θα έρθουν και οι επίτροποι. Oh, yeah. well, uh... on the topic. Energy efficiency and Brexit. Mr. Uh, Pocher report. Για την έκθεση του κυρίου Πόχε. Δίνω το λόγο σε άλλο συνάδελφο. Ε, συγγνώμη, ήμουν και στην Επιτροπή Μεταφορών και έπρεπε να τοποθετηθώ εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας για το Brexit σε ό,τι αφορά το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και της σχετικής οδηγίας και την πιθανότητα να μην υπάρξει συμφωνία ή ε, ε, και να υπάρξει συμφωνία με, το, με τη Μεγάλη Βρετανία. Σε σχέση με το θέμα αυτό, θέλω απλώς να παρακαλέσω όλους τους εμπλεκόμενους, όλους τους συνομιλητές μας να ε, το θέμα και οι τροπολογίες μας η έκθεσή μας να αφορά μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά, τεχνικά στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν ε, ε, να, πρέπει, να ζητάμε από τα κράτη-μέλη να προσφέρουν ακόμα περισσότερα όσον αφορά το ενεργειακό κόστος. Ε, ας μην προχωρούμε λοιπόν σε πολιτικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις, ας περιοριστούμε και ας αρκεστούμε μόνο στα τεχνικά, στα αριθμητικά στοιχεία, καθαρά, και μέσω αυτών να υπάρξει μια η αναγκαία προσαρμογή όσον αφορά τον επιμερισμό των ευθυνών και να εξασφαλίσουμε βεβαίω ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα δημιουργήσει ούτε ωφέλη αλλά ούτε και ιδιαίτερα βάρη σε επιμέρου χώρε. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, για την παρατήρηση αυτή. Θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μας. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι καταφέρατε να παραστείτε σήμερα εδώ. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές συνεδριάσεις πάρα πολλών επιτροπών και δεν μπορεί ένας ευρωβουλευτής να είναι σε 100 μέρη ταυτόχρονα. Γι' αυτό και είχαμε κάποιες απώλειες εδώ σήμερα στην Επιτροπή Ήτρε, αλλά παρόλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ. Βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει ζητήσει το λόγο για το θέμα αυτό. Οπότε να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο. Στις 9 το βράδυ. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα γίνει συνεδρίαση της δικής μας επιτροπής τουλάχιστον στο Στρασβούργο, αλλά θα γίνει συνεδρίαση, όπως είπα, στις 14 Ιανουαρίου. Είναι λίγος ο χρόνος, ε, βαίνουμε προς το τέλος της θητείας, οπότε καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι κάπως πιεστικά. Λοιπόν, για μισή ώρα θα είναι αυτή η συνεδρίαση, σας παρακαλώ να είστε εκεί.